Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Προηγουμένως όμως ε, δύο διαδικαστικά να αναγγείλω. Να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Τόγια. Mrs. she's not there. η κυρία Τόγια. Άρα η κυρία Καρδίνη η επόμενη.